για το πολιετές σχέδιο για τα αποθέματα βακαλάου, ρέγγας και άλλων ειδών στην Βαλτική. Τον λόγο έχει η κυρία Επίτροπος. Thank you very much, Madam President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, ο Επίτροπος Καρμένο Βέλε που είναι ε, ε, αρμόδιος ε, για το θέμα δεν παρευρίσκεται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τους κοιόδης εισηγητές και όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν τόσο να καταλήξουμε συμφωνία για το πολιετές σχέδιο για τη διαχείριση του αποθέματος του γάδου Ρέγκας και Σαρδελό στη Βαλτική θάλασσα. Το βαλτικό σχέδιο αυτό, το σχέδιο μάλλον της Βαλτικής θάλασσας ανήκει σε μια νέα γενιά πολιετές των ε, προγραμμάτων ε, πολύ σημαντικά εργαλεία για την ε, εφαρμογή της, πολιτι... της κοινής αλλιευτικής μας πολιτικής και για την υλοποίηση του πλέον σημαντικού στοιχείου για την καταπολέμηση της απόρριψης των ηχθείων των αλλιευμάτων. Ε, επιδιώκουμε μια πιο αποκεντρωμένη, ε, δηλαδή μια περιφερειακή διαχείριση. Θα ήθελα επίσης ε, να δράξω την ευκαιρία ούτως ώστε να κάνω και μια δήλωση σε σχέση με την περιφερειακή συνεργασία κατά την έγκριση, κατά εξουσιοδότηση πράξεων για τις διατάξεις περιφερειακού ελέγχου αυτού του προγράμματος. Θα εφαρμόσουμε το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού και την πρακτική που προβλέπεται στον βασικό κανονισμού σε σχέση με την περιφερειοποίηση των διαδικασιών. Θα συνεχίσει όπως ε, ε, ξεκίνησε το 2014. Είναι η αποκορύφωση μιας διαδικασίας ε, όπου συνεργάζονται διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς για να καταλήξουν σε συνενετικές λύσεις. Αυτή η διαδικασία καλύπτει τη βιομηχανία, τα Υπουργεία Αλληλείας των ενδιαφερόμενων χωρών, των συνομοθετών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Ε, καταλήξαμε σε μια ισορροπία και λάβαμε υπόψη τα βασικά αιτήματα των εμπλεκομένων φορέων. Ε, οι συνομοθέτες ε, επέτρεψαν με την συγκατάθεσή τους την έγκριση αυτού του πολιετού σχεδίου που έχει ιδιαίτερη σημασία και για άλλες περιοχές όπου θα καταστεί πλέον δυνατή μακροπρόθεσμη διαχείριση των αποθέσεων αλλιευτικών αποθεμάτων. Ε, θα υποβάλουμε λοιπόν προς εξέταση το έγγραφο για, τη νέα, για το νέο αυτό πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε. Ε, κύριος Βαλέσα, ε, δύο λεπτά. Thank you, Madam Chair. Ε, thank you, uh, Madam... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε. Αυτό το πρώτο σχέδιο διαχείρισης της αλίας υπό τη νέα CFP είναι αποτέλεσμα σκληρού αγώνα μετά από δυσχερείς και μακρές διαπραγματεύσεις όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπίθη να κάνει πολλές παραχωρήσεις. Περιλάβαμε διατάξεις που πιστεύουμε ότι θα είναι επαρκής για την διάσωση των αποθεμάτων αυτών. Πρέπει να τεθεί σε ισχύ το δυνατόν συντομότερο το νέο αυτό σχέδιο για να διασώσει τα αποθέματα για το 2017. Είναι αναγκαίο να δράσουν με υπεύθυνο τρόπο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να δείξουν ότι τηρούν τις βασικές αυτές αρχές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε τη δέσμευσή του υπέρ αηφόρων ε, αλληλευτικών αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οφείλω να ζητήσω το ίδιο να κάνουν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο ερωτήσει. Οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επόμενα χρόνια για το συνολικό επιτρεπόμενο απόθεμα για τον Βακαλάο θα βασιστούν στι ίδιε επιστημονικέ συμβουλέ και στου κανόνε που περιλαμβάνει το νέο αυτό σχέδιο διαχείριση. Υπάρχει κάποιο σενάριο όπου οι κανόνες που απορρέουν από το σχέδιο αυτό να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι κρίσιμο να χρησιμοποιηθούν, να εφαρμοστούν δηλαδή οι νέοι αυτοί κανόνες ταχύτατα, διότι οι επιστημονικές συμβουλές μας οδηγούν σε πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Τα αλληλευτικά αυτά αποθέματα βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Τα αποτελέσματα της αποτυχίας να εφαρμοστούν οι κανόνες έως τώρα έχουν οδηγήσει τους επιστήμονες να μας λένε ότι πρέπει λίγο πολύ να κλείσει η αλία αυτή. Ευτυχώς το νέο διαχειριστικό σχέδιο για την Βαλτική έχει νέους κανόνες καθώς και κάποιες ρήτρε προφύλαξη. Μετά από 10 μήνε δύσκολων διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι διαπραγματεύσει αυτέ μα προσφέρουν επιτέλου ένα σχέδιο το οποίο διατηρεί του ε, στόχου του βασικού κανονισμού για να εξασφαλιστεί ότι η αλευτική δραστηριότητα στην Βαλτική θα γίνεται με τρόπο βιώσιμο, αηφόρο και οικονομικά αποδοτικό, που δεν θα επιβαρύνει με περιττό τρόπο το περιβάλλον. Πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ρόντουστ. 2 και 30 εκ της ε, Σοσιαλιστικής και Δημοκρατικής Ομάδος. Ήταν πράγματι εντατικές και μακρότατες οι διαπραγματεύσεις αυτές. Αύριο πρόκειται να ψηφιστεί το κείμενο για το πρώτο πολιετές σχέδιο στην βάση της νέας αναθεωρημένης κοινή αλληλευτικής πολιτικής και πέρασε μέσα από, τρεις, μέσα από 8 τριμερείς διαλόγους. Χρειάστηκε πολλή ενέργεια για να ηρεμήσουν τα νερά μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που θα μας είχαν πνίξει αν δεν τα είχαμε μπορέσει να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Βαρέλνσα για την εργασία του και για τον τρόπο προσεγγίσεως που οδήγησε στο ότι οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απηχούνται επαρκώς στο κείμενο. Τα τρία θεσμικά όργανα πέρασαν από διαπραγματεύσεις διαρκείας 10 μηνών και δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε όλα τα θέματα και ιδίως για την διατηρησιμότητα των αποθεμάτων. Όμως οι διατάξεις του βασικού κανονισμού πρέπει να εφαρμοστούν. Το Συμβούλιο δεν το δεχόταν αυτό και επέμεινε να υπάρξει κάποια ευελιξία. Στο τέλος καταλήξαμε σε συμβασμό. Σε ό,τι αφορά τις βασικές αξίες, τις βασικές τιμές για τη θνησιμότητα των αποθεμάτων, τα βρήκαμε με το Συμβούλιο. Η ευελιξία δίνεται αλλά με κάποιους όρους. Μετά από θετική ψηφοφορία, την οποία αναμένω αύριο, θα πρέπει από τη δική μας σκοπιά το νέο αυτό πολιτές σχέδιο για την, <clears throat> να αρχίσει να εφαρμόζεται ήδη από τον Οκτώβριο για, για τον καθορισμό των ανώτατων επιτρεπόμενων αλλιευμάτων. Πρέπει να κάνει τα απαραίτητα το Συμβούλιο έτσι ώστε να δημοσιευτεί το αργότερο τον Αύγουστο στην, στο επίσημο έντυπο της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως το νομοθέτημα. Τα είδη τα οποία αναφέρονται στον τίτλο του κανονισμού τα, αποθεμάτα του, δηλαδή βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Το ίδιο και οι αλλοί. Πρέπει να ληφθούν τα μέτρα αυτά λοιπόν ταχύτατα. Εν ώψη της καταστάσεως αυτής στην Βαλτική χαίρομαι που μπορούμε μέσω του σχεδίου να προσφέρουμε και υποστήριξη μέσω του Ταμείου της Θάλασσας. Εγώ θεωρώ το σχέδιο αυτό ως ένα βασικό σχέδιο για την περαιτέρω πορεία μιας αηφόρου αναπτύξεως στην Αλία. Χαίρομαι που στα κείμενα αυτά βάζουμε ασφαλή όρια τα οποία οφείλουν να τηρήσουν οι Υπουργοί Αλίας διότι εξασφαλίζουν αυτά τα σχέδια και αυτές οι τιμές την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και αποτελούν εγγύηση για την βιωσιμότητα και την αηφορία. Αποτελεί το σχέδιο αυτό ένα σημαντικό βήμα και χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ. κύριε ο κύριος Ότς, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης για αυτά τα είδη ψαριών είναι πολύ ε, σημαντικό και είναι αποτελεσματικό. Είναι το πρώτο τέτοιο είδου σχέδιο που έχει αναπτυχθεί μέσω της νέας αλληλευτική πολιτικής. Πρόκειται για, μια, ε, για τη διαχείριση διαφόρων ειδών που λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση των ειδών μεταξύ του. Είναι καλό αυτό γιατί ξέρουμε ότι η βιοποικιλότητα στην Βαλτική πρέπει να να αποκατασταθεί και η διαχείρισή της να βασιστεί σε μια ισορροπημένη προσόγηση και σε ε, στα, στέρεα επιστημονική γνώση. Κάποιες παρατηρήσεις από πλευρά μου θα πρέπει να είναι περιφερειακή προσέγγιση και βέβαια κάποιες περιοχές θα πρέπει να είναι κλειστές στην αλληλεία για να προστατευτούν τα οι αλληλευτικοί πόροι. Επίσης η αλληλεία θα μπορούσε να απαγορεύεται για κάποιες περιόδους εφόσον υπάρχουν ε, ε, λόγοι γι' αυτό. Ε, περιορισμός της βιομηχανικής αλληλείας. Επίσης και αν ε, στην Πολωνία πρέπει να κατασκευαστούν αιωλικά πάρκα ε, ε, στη Βαλτική θα πρέπει αυτό να γίνει εκεί όπου δεν γίνεται αλληλεία. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για την καλή έκθεση. Για δύο, λεπτά ο κύριος Πρόεδρε Επιτροπέ. Ε, θεωρούσαμε ότι θα ήταν απλά τα πράγματα, τελικά ήταν πολύ δύσκολες ε, οι διαπραγματεύσεις. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να, να ευχαριστήσω όλος ιδιαίτερα ε, τον κύριο Βαλέσα για τις προσπάθειές του, διότι πραγματικά εισάκουσε τις επιθυμίες μας και κατέληξε σε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ουλρή και Ρόντουστ, χωρίς τις προσπάθειές της δεν θα είχαμε καταλήξει σε αυτό το αποτέλεσμα που είναι τόσο σημαντικό για την αλληλευτική πολιτική και ε, πραγματικά ε, κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων διαπραγματεύσεων με στηρίξατε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εγκάρδια. Γιατί ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, ε, διότι είναι κλειστή η θάλασσα, κλειστή η θάλασσα η Βαλτική, είναι μολυσμένη σε σχέση με αντίστοιχες θάλασσες ε, έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και επίσης ε, υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συμφέροντα των παρακτήων χωρών. Και φυσικά ξέρουν όλοι ότι το βάπτισμα του πυρός είναι κάτι δύσκολο και επειδή πρόκειται για το σχέδιο μια νέας γενιάς ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Ε, επίσης άλλη δυσκολία είναι ότι δεν ακολουθούν τις οδηγίες μας και τους κανονισμούς μας τα ψάρια στη συμπεριφορά τους και στην αναπαραγωγή τους. Ε, Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, ε, επίσης να αντικατασταθούν αλληλευτικές δραστηριότητες διότι δεν υπάρχουν άλλες δραστηριότητες σε πολλές τέτοιες ε, παράκτιες χώρες. Ξέρουμε επίσης ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις διότι υπήρχαν και άλλα συμφέροντα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε στόχο που επιδιώκαμε, αλλά το καταφέραμε και πάλι σας ευχαριστούμε κυρία Ρόντος. Ευχαριστούμε κύριε Τόρβελς, ε, κυρία Χάζεκαμπ ε, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κανείς, ε, πιστεύω εγώ, δεν μπορεί να δηλώσει ικανοποιημένο με αυτό το σε σχέδιο διαχείριση του αποθέματος για την Βαλτική θάλασσα, ούτε οι ούτε και τα ψάρια. Ε, διότι μιλάμε για την, ε, τον δίκτυ FMSY, μέγιστη βιώσιμη απόδοση αλληλείας ε, και τελικά όμως οδηγούμαστε σε υπεραλίευση, δηλαδή ε, αυτά τα αποθέματα υπεραλλιεύονται στο μέγιστο και δεν μιλάμε για πράγματα, μιλάμε για ε, όντα. Δεν αρκεί το να ορίζουμε ανώτατα όρια αλίευσης ε, και πέρα από αυτό μέσα στο σχέδιο ε, μιλάμε για την μέγιστη βιώσιμη απόδοση χωρίς να ορίζουμε όμως ε, τι εστί υπεραλίευση και τελικά αποδυναμώνουμε την κοινή αλλιευτική πολιτική. Πιστεύω ότι θα ανοίξει αυτό την πόρτα, την κερκόπορτα και για άλλες θάλασσες όπως η Βόρεια Θάλασσα. Πολύ αντισταθήκατε ε, σε αυτό το σχέδιο πολυετούς προγράμματος ε, και οι συγκητές θα θέλουν να πιούμε και σαμπάνι για να το γιορτάσουμε μετά την αυριανή ψηφοφορία. Πραγματικά θέλετε να το γιορτάσετε εάν ε, μεταφράζεται έτσι η φιλοδοξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. το αποτέλεσμα είναι ότι θα αδειάσουν οι θάλασσε και ε, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό κατά τη διάρκεια τη δική μα ζωή η κυρία Έγκστρομ. ειδου προγραμματα δυο λεπτα η Πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαλέσα και την δουλειά που έκανε και τη βοήθειά του για να καταλήξουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι το πρώτο πρόγραμμα διαχείριση στο οποίο κατέληξαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πόσο μπορούμε να ψαρεύουμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολε οι διαπραγματεύσει και καταφέραμε καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία να υποστηρίξουμε την θέση του Κοινοβουλίου, δηλαδή ε, διακοπή τη ε, υπεραλίευση. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε όλους τους παράγοντες μέσα σε τέτοιες θάλασσες, κυρίως στις κλειστές θάλασσες. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο αυτό. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε περιθώρια ασφάλειας όταν ε, διαπραγματευόμαστε τις μέγιστες ε, βιώσιμες αποδόσεις ε, αλίες. Για να έχουμε ζωντανά αλλιευτικά αποθέματα. Δεν μπορούμε διαρκώς να αλλιεύουμε μέχρι τα ανώτατα όρια. Θα πρέπει να επιδιώξουμε χαμηλότερα όρια για να μπορέσει να αναπληρωθεί το απόθεμα. Αντί να μιλάμε για το FMSY, θα πρέπει να δούμε ε, ε, ε, ότι τα κράτη μέλη αυτό που τους ενδιαφέρει να κάνουν είναι να ψαρεύουν κοντά στο επίπεδο FMSY ή υπέρ αυτού. Το αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε ανταυτού και τον βασικό κανονισμό και τους αρχικούς στόχους κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Έρχεται και η πρώτη δοκιμή. Λάβαμε ιδιαίτερα ανησυχητικέ εκθέσεις την περασμένη εβδομάδα για την κατάρρευση των αποθεμάτων γάδους στην Βαλτική. Ε, ο Επίτροπος Βελέ θα πρέπει να λάβει υπόψη ε, αυτές τις μελέτες ε, και πώς βάσει αυτού του προγράμματος θα προστατεύσουμε τα αλλιευτικά αποθέματα διότι περιγράφονται προστατευτικά μέτρα όμως δεν μεταφράζονται στα όρια, στα βιώσιμα όρια αλλιεύσης. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόζουμε τις αποφάσεις που λαμβάνουμε και όχι ε, να τις ε, αδειάζουμε από το περιεχόμενό τους. Είναι υποκρισία. Ε, υπονομεύουμε την ίδια την αλληλευτική πολιτική και την ευρωπαϊκή συνεργασία μη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις μας. Ευχαριστούμε κύριος Μάτο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, απέναντι σε δια... ενώπιον διαφόρων καταστροφολογικών ε, εισηγήσεων που ακούσαμε, εγώ πιστεύω πως φέτος ε, δίνουμε ένα μέτρο για να μπορέσουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσουμε τους ελευθερικούς μας πόρους. Αυτό που συζητάμε σήμερα όχι μόνο εξασφαλίζει ένα πολιετές ε, σχέδιο ε, διαχείρισης των αλληλευτικών αποθεμάτων στις θάλασσες της Βόρειας Ευρώπης για το, τόνο, τη Ρέγκα και την ε, Σαρδελόρεγκα ε, αλλά επίσης βλέπουμε επιστημονικές αποδείξεις για όλα αυτά. Θα πρέπει να μιλήσουμε κυρίως όμως για αρμοδιότητες και εγώ θέλω να τονίσω την αρμοδιότητα που έχει κάθε ένα από τα θεσμικά όργανα και θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Ο στόχος λοιπόν είναι να θεσπιστούν πολιετή προγράμματα τα οποία αναλαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές ε, που αφορούν τη διαχείριση αυτή της αλληλευτικής δραστηριότητα ε, με εγγύηση όμως για μια βιώσιμη εκμετάλλευση τη ε, αλληλεία και προστατεύοντας τη δραστηριότητα των αλληλεών μα Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σα ευχαριστώ. 1,5 λεπτό Σεράου Σάντος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ το εισηγητή που είχαμε εδώ, τους εισηγητές Βαλέσα Ρόντουστ και σίγουρα τους κοιόδης εισηγητές που πολλούς μήνες προσπάθησαν ώστε η θέση του Ευρωκοινοβουλίου να είναι όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτική του σώματος. Υπάρχουν κάποιες επίμαχες τροπολογίες Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτή η λύση θα μπορέσει να συμβάλλει στην διατήρηση των ειδών ε, σε επίπεδα βιομάζας που θα επιτρέψουν την βιώσιμη εκμετάλλευσή τους. Ε, θα μπορέσουμε να, έτσι, να αποκαταστήσουμε τις περιοχές αυτές. Όμως θα πρέπει και διαρκώς να επαληθεύουμε αν είναι αν όλα αυτά είναι προσαρμοσμένα με τη νέα αλληλευτική πολιτική. Πέρα από αυτά τα θετικά βήματα θα πρέπει να τονίσουμε και το τι συμβαίνει στην ε, Μεσόγειο. Πολλές ε, αλληλευτικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υγιείς. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την αντοχή των οικοτόπων και των διατροφικών αλυσιδών των διαφόρων ειδών και γι' αυτό θα πρέπει να, εισαχθούν, να, να οριστούν συγκεκριμένες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές αλλά και ποσοστώσεις αλλά και μια προληπτική πολιτική που να μπορεί να ε, αντιπαρέλθει στα, αρνητικέ αρνητικές επιπτώσεις της αλίας. Ευχαριστώ. Βαντάλεν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, φτάσαμε επιτέλους σε μια συμφωνία για την Βαλτική με αυτό το σχέδιο που το οποίο παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο και μετά 1,5 χρόνο μετά έχουμε μια νομοθετική συμφωνία. Μακρύς δρόμος, πολυετές σχέδιο, το οποίο ε, μάλιστα απασχόλησε αρκετό καιρό το Κοινοβούλιο. Δηλαδή ρωτώ α, τι συμβαίνει με άλλα πολυετή προγράμματα. Ίσως θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε τα πράγματα στο μέλλον, γιατί το πλαίσιο είναι σαφές. Έχουμε επιλέξει συγκεκριμένες περιοχές, μέσα στις, μάλλον κάποια φάσματα, εντός των οποίων μπορούν να εφαρμοστούν ποσοστώσεις. Και αυτό είναι απαραίτητο γιατί υπάρχει ανάμεκτη αλληλεία σε αυτές τις περιοχές και μπορεί να επιτευχθεί μια μέγιστη βιώσιμη αλληλεία και όλα αυτά τα στόκ να να ωφεληθούν. Είναι διπλός ο στόχος λοιπόν για την κοινή ελευτική πολιτική. Τέλος, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαλέσα και την ομάδα του για την εξαιρετική τους, ε, τα, εξαιρετικά τους αποτελέσματα στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Μπιλμπάου. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Βαλέσα και την διαπραγματευτική ομάδα για την ε, προσήλωσή του σε αυτό το πολιετές πρόγραμμα για το τόνο, τη Ρέγκα και τη Σαρδελόρεγκα στην Βαλτική. Και ελπίζω ότι η διαφάνεια αυτή θα επιτρέψει και τον ορισμό των αληφτικών ποσοστώσεων. Η αντίσταση του Συμβουλίου, παρότι το Κοινοβούλιο έχει δυνατότητα συναπόφαση σε αυτή την περίπτωση, εμποδίζει ε, την επίλυση των προβλημάτων για άλλα είδη όπως ε, το σαφρίδι και, το, και ο μερλούκιος. Ε, εδώ θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός των ποσοστώσεων όμως με μεθόδους όχι συμβατές με την ανταγωνιστικότητα την οποία εμείς υποστηρίζουμε αλλά και την μεταρρύθμιση στην αλληλεία. Οι αλληλείς είναι θύματα και γι' αυτό είμαστε υπέρ στην, της γενίκευσης αυτού του συστήματος προγράμματα διαχείρισης δηλαδή πολυετή που πράγμα που είναι καλύτερο για την θάλασσα και την ισορροπία της και για όσους ζουν και αλλιεύουν σε αυτήν, στη θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, Μαρτίνες, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Είναι πρόοδο το ότι αναλύουμε την κατάσταση της αλληλείας στη Βαλτική με ε, τρόπο κοινό για διάφορα είδη, γιατί αυτό βοηθά στη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και να φροντίσουμε ώστε αυτές οι νομοθεσίες να αντιστοιχούν στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και περιφέρειας. Οι ανάγκες των αλλιέων δεν λαμβάνονται πάντοτε υπόψη από την Ένωση. Οι αλλοί μας και ιδιαίτερα αυτοί που αλλιεύουν ε, ε, είδη τα οποία είναι ήδη λιγοστά ε, κινδυνεύουν. Πρέπει να σεβαστούμε τη ζωή τους και την κουλτούρα τους. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε χωρίς να ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους ώστε να έχουν και αυτοί ένα μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ώστε να υπάρχει βιώσιμο πρότυπο εντός των κρατών και να επαγρυπνούμε όσον αφορά τα είδη για να μην, να μην επιτρέψουμε τα μεγάλα αλλιευτικά σκάφη τα οποία αλλιεύουν δίπλα στους ε, βιοτέχνες ε, ψαράδες ε, να καταστρέψουν τα αλλιευτικούς σπόρους. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό κούνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ <clears throat> και όλους τους συναδέλφους που συμμετέσχουν στις διαπραγματεύσεις για την επιμονή τους και για την επιτυχή λύση που έδωσαν στο πρόβλημα των αποθεμάτων, των λευτικών αποθεμάτων δηλαδή, για την Βαλτική που εξασφαλίζει ασφάλεια στους αλληλείς και τη δυνατότητα οικονομικών αποζημιώσεων. Και το FMSY, δηλαδή η ελάχιστη, η μέγιστη βιώσιμη απόδοση, δίνει και μια ανάσα στη, στα αλλιεύματα για μια περίοδο 6, 7, 10 ετών και επιτρέπει με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, δηλαδή ανάλογα με την αναπαραγωγική δυνατότητα των αδειγμάτων, να μπορέσουν να έχουν μια ένα ασφαλή σχεδιασμό και οι Από την άλλη μεριά χαίρομαι για το γεγονός ότι άλλαξαν, τροποποιήθηκαν ορισμένα πράγματα, τα οποία θα συνεπέφεραν μια σημαντική γραφειοκρατική επιβάρυνση, τη κατάργηση δηλαδή των ημερών στην θάλασσα, ε, ορισμένα άλλα επίσης και στην περίπτωση που δένουν τα σκάφη να δίνεται μια οικονομική αποζημίωση στους αντίς. Ευχαριστούμε. Μαρίνιο Εμπίντο για ένα λεπτό επίση. Ε, τελευταία φορά που εγκρίναμε τέτοιο πρόγραμμα ήταν το 2008. Ε, ε, συγχαρητήρια για το νέο πρόγραμμα, συγχαρητήρια προς τους, ε, προς τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως έπρεπε να είναι πιο φιλόδοξη στην πρότασή της, διότι αυτό που διακυβεύεται είναι τα αυθύνοντα αλλιεύματα αυτών των τριών ειδών της ρέγκας, της αρδελόρικας και του βακαλάου. Ε, θα πρέπει να μεριμνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία όλων των ελευθερικών αποθεμάτων αλλά και του θαλασσίου περιβάλλοντος ε, διότι μόνο έτσι θα μπορέσει να εκπληρωθεί ο πρώτος και βασικός στόχος της κοινή αλιευτικής πολιτικής αυτή η μέγιστη δηλαδή βιώσιμη απόδοση αλίας για μια χώρα όπως η Πορτογαλία όπου ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει από τη θάλασσα κυρίως μιλώ για τους αλίες όλα τα μέτρα που συμβάλλουν στην προστασία ε, ε, της, ε, του θαλασσίου περιβάλλοντος είναι ευπρόσδεκτα. Ευχαριστούμε κύριο Σόλτς. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με το πολιτές σχέδιο για την Βαλτική λαμβάνουν επιτέλους οι αλλοίς και στη δική μου εκλογική περιφέρεια, το Μέκλεν Βουφό, Απόμενη και το Σλέζι Χολστάιν, την απαραίτητη ασφάλεια σχεδιασμού πρόκειται για μια δυνατότητα που τους δίνεται να σχεδιάσουν την αλία με τρόπο βιώσιμο. Ως αριστερά είμαστε απολύτως υπέρ διότι διασφαλίζονται σταθερές ποσότητες αλλιευμάτων και επομένω μια σταθερή βάση εισοδήματο για τους αλείς. Το Διεθνές Συμβούλιο Θαλασσίων Ερευνών προτείνει μείωση των, των ε, ε, αλλιευσίμων ποσοτήτων για τον γάδο της τάξης του 85% στην Δυτική Βαλτική πάβει επιτέλους μια πράξη, στη, μια πρακτική μάλλον, η οποία επέτρεπε να ορίζονται τα όρια των αλλιευμάτων και ακόμα και αντίθετα με τις επιστημονικές συμβουλές. Τώρα πλέον θα ισχύει η αρχή ότι αλλιεύεται μόνο η ποσότητα αλλιεύματος που μπορεί να αναπαραχθεί. Όπως είναι τώρα, το πολιετές σχέδιο προβλέπει και δυνατότητες στήριξης των αλλιέων και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί ταχύτατα και με τρόπο ευθύ και μη γραφειοκρατικό. Θα αρχίσει η διαδικασία Catch the Eye. Τρεις παρεμβάσεις έχουμε. Κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Συμφωνία Πολιτής για τη Βαλτική δημιουργεί τη βάση για μια βιώσιμη αλληλεία στα πολύ μεγάλα αποθέματα της Βαλτικής θάλασσας. Είναι το πρώτο τέτοιο είδους σχέδιο μετά από τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και πιστεύω πως αυτό το σχέδιο είναι συνεκτικό και σύμμορφο με τις αρχές της μεταρρύθμισης. Υπογραμμίζω την σημασία του να εγγυηθούμε ότι η διαχείριση των στόκ στη Βαλτική θάλασσα θα πρέπει να βασίζεται σε ε, ε, επιστημονικά στοιχεία. Θα πρέπει εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα την περιοχή, να δουν αν μπορούν να, να προσαρμόσουν τα μέτρα στην ιδιαιτερότητα τη αλληλευτικής δραστηριότητα. Η εν λόγω ε, συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την επεξεργασία ανάλογων πολιετών ε, προγραμμάτων με το ίδιο μοντέλο για την αλληλεία σε άλλε γεωγραφικέ ε, περιοχέ. Τα πολιετή προγράμματα διαχείρισης φάνηκαν χρήσιμα για τη βιώσιμη διαχείριση των αλληλευτικών πόρων γιατί θεσπίζουν ξεκάθαρους κανόνε για τη διαχείριση των στόχων ΠΑΣΟΚ, η αρχή της μέγιστης βιώσιμης απόδυσης εγγυάται συνθήκες σταθερότητας και προβλεψιμότητας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριος Μαριάς. Ε, η Ολλανδική Προεδρία κατέληξε στις 15 Μαρτίου του 2016 σε μια προσωρινή συμφωνία με την οποία επιδιώκεται η θέσπιση πολιετού σχεδίου για την αλία βακαλάου ρέγκα και σαρδελόρεγκα που αποτελούν σημαντικά είδη στη βαλτική θάλασσα. Ωστόσο, σύμφωνα με γνωμοδοτήσει του Διεθνού Συμβουλίου για την Εξερεύνηση τη Θάλασσα, οι σημερινοί ρυθμοί εκμετάλλευση ορισμένων αποθεμάτων δεν συνάδουν με την επίτευξη μέγιστη βιώσιμη ανάπτυξη. Επομένω, είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει άμεσα μέτρα, ώστε τα αποθέματα αυτών των τριών ειδών στη Βαλτική να αλλιεύονται σύμφωνα με την αρχή τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ταυτόχρονα όμω, κυρία Μπιενκόφσκα, κυρία Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κοιτάξει και στον Νότο και να λάβει μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των ελλήνων αλλιέων που έχουν φτωχοποιηθεί από την τρόικα και τα μνημόνια. Σας μεταφέρω κυρία Μπιενκόφσκα την κραυγή διαμαρτυρίας των Ελλήνων αλλιέων που δεν αντέχουν άλλο την φόρο επιδρομή της Τρόικας, τη διάλυση του πρωτογενού τομέα και τη μερκελική λιτότητα. Ευχαριστώ. Ε, συνήθως, έτσι, ναι, λέει η Πρόεδρος, το γνωστό, η γνωστή τριάδα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους συναδέλφους. Μετά από 8 τριμερείς διαλόγους κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σε αυτό το πολιετές σχέδιο για τη διαχείριση των αποθεμάτων ε, γάδου Ρέγκας και Σανδελόρεκα στη Βαλτική. Είναι κλειστή η θάλασσα η Βαλτική και χρειαζόμαστε πολυετή προγράμματα διαχείρισης των αποθεμάτων. Όμως θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Ε, είναι επιτακτική ανάγκη η ύπαρξη ενός συγκρίσιμου προγράμματος διαχείρισης για την Αδριατική ε, θάλασσα. Το χρειαζόμαστε το ταχύτερο δυνατόν. Κάποιοι είπαν πως θα έπρεπε να απαγορευτεί η αλία κάποιων ειδών στη Βαλτική και ενδεχομένως να είναι πολύ αργά ήδη για κάποια είδη στην Αδριατική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει να εξετάζει αυτό το θέμα ε, ε, μέτρα συντήρησης των αποθεμάτων, διατήρηση συγγνώμη, των αποθεμάτων για την Αδριατική. Ε, η κυρία Μπιενκόσκα θα απαντήσει εξ ονόματος τη Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις τους και φυσικά θα διαβιβάσω τις ε, πληροφορίες και τις ερωτήσεις στον Επίτροπο Βέλα και θα λάβετε λεπτομερείς απαντήσεις. Θα ήθελα όμως ε, εν συντομία να σχολιάσω δύο σημεία. Πρώτον, θα ήθελα να τονίσω ότι το πολιετές σχέδιο για τη Βαλτική είναι το πρώτο μιας νέας γενιάς ε, διαχειριστικών προγραμμάτων και όταν θα καταθέσουμε τις επόμενες προτάσεις για, τα, για την αλία σύντομα και όσο γνωρίζετε αυτό είναι και νομική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, διότι πρέπει να συμμορφωθεί με τις ε, τρέχουσες υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις ε, θα πρέπει να ξέρετε ότι να λάβετε υπόψη μάλλον ότι τέλη Αυγούστου, αρχέ Σεπτεμβρίου θα έχουν καταδεθεί οι προτάσει, ώστε εγκαίρω να ε, προληφθεί το έδαφο για τι συζητήσει στο Συμβούλιο τον ε, Οκτώβριο. Αν έχει τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο, μέχρι τώρα και τώρα είναι ε, κοινή η ευθύνη των δύο συνομοθετών για την εφαρμογή του προγράμματο, τότε η νέα πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βασιστεί σε αυτό το νέο πολιετέ πρόγραμμα. Έτσι, ελπίζω να οργανώσετε την επίσημη τελετή υπογραφή σε σύντομα ε, για να τεθεί και σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατόν. Ε, επίσης να το προσθέσω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τις εφιστάμενες διατάξεις για τις δικλείδες ασφαλείας ε, και τις ε, υπόλοιπε διατάξεις που υπάρχουν στην νομοθεσία για να καταθέσει τα νέα προγράμματα. Αυτά προς το παρόν και σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε και ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση.